συζήτηση αυτή. Εξ ονόματος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταρχάς έχει το λόγο ο Επιτρόπος Μίμητσα. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Καλωσορίζω την ευκαιρία της κατεπίγουσας ε, συζητήσεως για την εκτέλεση των 8 φυλακισμένων στην Ινδονησία. Κάτι που απογοήτευσε και έθλιψε ε, και εμάς και την διεθνή κοινότητα Είμαι σίγουρος ότι τα αξιότιμα μέλη μοιράζονται μαζί μας την έκφραση της βαθιάς απογοητεύσεως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρή θέση καταρχήν κατά της θανατικής ποινής σε όλες τις περιπτώσεις και περιστάσεις και εργάζεται προς την κατάργηση της ποινή, της θανατικής σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα στόχος και προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής όσον αφορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εξωτερική πολιτική είναι προφανή η υποχρεώσει που έχουμε αναλάβει στι κατευθύνσει γραμμέ για τη θανατική ποινή τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Οι πρώτε κατευθυντήριε γραμμέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υθετήθηκαν από το Συμβούλιο το 1988 και αναθεωρήθηκαν ακολούθως και πλέον προσφάτω το 2013. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φρονεί ότι η θανατική ποινή είναι απάνθρωπη και βίαιη και πουθενά δεν έδειξε ότι μπορεί να αποτρέψει την διάπραξη εγκλημάτων. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η κατάρριξη ανατικής ποινή είναι κάτι ουσιαστικό για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για την προοδιακή ε, ανάπτυξη και εξάπλωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδήποτε λάθο τη δικαιοσύνη, κάτι που είναι αναπόφευκτο σε οποιοδήποτε νομικό σύστημα, είναι κάτι αμετάκλητο για αυτή την Οι πρόσφατες αυτές εκτελέσεις είναι ιδιαίτερα ε, εξωφρενικές, διότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ τα αδικήματα που αφορούν τα ναρκωτικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό του σοβαρού εγκλήματος. Μέσω της εξωτερικής πολιτικής η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στις παγκόσμιες προσπάθειες για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Από το 1993 μέχρι το 2012 ο αριθμός των χωρών που κατήργησαν την θανατική ποινή δια νόμου για όλα τα εγκλήματα ανέβηκαν από 55 σε 97 από το Δεκέμβριο του 2012, 140 χώρες, πάνω από τα 2 τρίτα των χωρών του κόσμου, είχαν καταργήσει στην πράξη ή διανόμου ε, τη θανατική ποινή. Δυστυχώ στην Ασία είναι ανάμεικτη εικόνα. Το Πακιστάν είναι το πιο πρόσφατο ανησυχητικό παράδειγμα, διότι παραβιάστηκε το πάγωμα, το μορατόριο και επανελήφθησαν οι εκτελέσεις τρομοκρατών εκτελέσεις που ήδη έχουν φτάσει τις 100 φέτος. Η ευρύτερη περιοχή έχει χώρες όπως η Κίνα, το Ιράκ, το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία που είναι στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίω όσον αφορά τις εκτελέσεις Ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των ασιατικών χωρών νόμιμα στο νόμο τους έχουν διατηρήσει τη θανατική ποινή. Πέντε ασιατικές χώρες έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή, το Μπουτάν, η Καμπότζη, το Νεπάλ, η Μογγολία και οι Φιλιππίνες. Αυτή η εικόνα με αντιθέσεις της περιοχής δείχνει ότι υπάρχουν κινήσεις όσον αφορά τον περιορισμό της ανετικής ποινής στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη και προς επανάληψη των εκτελέσεων στην Ινδία, την Ιδονησία, τη Μαλαισία, το Πακιστάν και το Βιετνάμ. Ή ενίσχυση της νομικής βάσης για τη θανατική ποινή όπως στο Μπρουνέ και στις Μαλδίβες. Η Ινδονησία ε, είναι επιτυχές παράδειγμα της μετάβασης προς τη δημοκρατία έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ασία. Η Ινδονησία είναι βασικός παίκτη και φορέας στην ΑΣΕΑΝ που έχει περίπου το 40% του ΑΕΠ και του πληθυσμού και είναι μεγάλος φορέας σε παγκόσμια κλίμακα και μέλος των G20 και είναι μία από τις τα, με, ταχύτερα αναπτυσσόμενες μέσες τάξεις εκεί όπως έχει και το μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό στον κόσμο. Η Ινδονησία έχει τον τέταρτο πληθυσμό στον κόσμο με 250 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο και είναι δημοκρατία, αλλά η δημοκρατία αυτή δεν μοιράζεται μαζί μας όλες τις αξίες μας. Η ηρωνία είναι ότι οι εκτελέσεις αυτές έγιναν με πολύ δημοκρατικό τρόπο σε μια χώρα που είναι από τις πιο ελεύθερες και δημοκρατικές της Νοτιοανατολικής Ασίας με ισχυρό και δραστήριο κοινοβούλιο ε, και κοινωνία των πολιτών πολύ ζωντανή ε, ήταν κάτι που δημιούργησε μεγάλη αγωνία στους φυλακισμένους και στις ε, οικογένειες διότι το όλο θέμα εκτελήχθηκε σε αργή κίνηση. Τώρα στρεφόμενος προς τις συγκεκριμένες μας δραστηριότητε. είπατε εκπρόσωπος προέβησε τρεις δηλώσεις εκφράζοντας βαθιά λύπη για την χρήση της θανατικής ποινής στην Ινδονησία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεργαστεί στενά με τα κράτη-μέλη ε, και που έχουν ε, δικούς τους υπηκόους που περιμένουν εκτέλεση. Καλέσαμε τις, ο πρόεδρος και την πρόεδρος καλέσαμε την, ε, τις αρχές της Ινδονησίας να σταματήσουν εκτελέσεις και να προχωρήσουν προς ένα οριστικό μορατόριο πάγωμα των εκτελέσεων. Οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουν χρησιμοποιήσει όλους τους διπλωματικούς τρόπους και μέσα για να θίξουν το θέμα της ανατικής ποινής με τους ομολόγους τους της Ινδονησίας. Προτιθέμεθα να ξεκινήσουμε σύντομα περιφερειακή εκστρατεία ευαισθητοποίησης με τίτλο «Απομακρυνόμενη από τη θανατική ποινή στην Ανατολική Ασία». Θα ηγηθεί η κοινωνία των πολιτών της περιοχής και άτομα και τοπικές οργανώσεις κοινωνια των πολιτών Γνωρίζω ότι αξιότιμα μέλη αυτού του Κοινοβουλίου ήταν δραστηρία και προσπάθησαν να πείσουν την Ινδονησιακή κυβέρνηση για την ανάγκη κατάργηση θανατικής ποινή και ε, έγιναν προσπάθειες και γίνονται για να σταματήσουν και άλλες εκτελέσεις. Αξιότιμα μέλη, σε παρεμβάσεις Έχουμε καταστήσει σαφές ότι σεβόμαστε την κυριαρχία της Ινδονησίας και προσφέρουμε και πολιτική υποστήριξη και πραστική αρρωγή για την καταπολύμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και άλλων δραστηριοτήτων εγκληματικών που δημιουργούν προβλήματα για την κοινωνία της Ινδονησίας και πέραν αυτής. Σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή με τις αρχές Ινδονησίας όσον αφορά την χρήση της θανατικής ποινής Προσβλέπω στο να ακούσω τις απόψεις των αξιοτήμων μελών και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Επιτροπή Μίμητσα και τώρα εξ ονόματος των ομάδων έχουμε του ομιλητές. Τρία λεπτά ο κύριος Ντάνζον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εδώ δεν είμαστε δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί δεν αποφασίζουμε για το κατά πόσο είναι ένοχοι ή αθώοι ή ύποπτοι που δικάζονται στην Ινδονησία. Είμαστε όμως πολιτικοί, εκλεγμένοι από τους πολίτες για να εκπροσωπήσουμε αξίες οι οποίες σήμερα μας επιβάλλουν. Να απαιτήσουμε από τις Ινδονησιακές αρχές οι πολίτες μας, όπως κάθε ύποπτος, να έχουν δικαίωμα σε δίκαιες δίκες που να σέβονται τα δικαιώματά τους, το δικαίωμά τους να υποστηρίξουν τον εαυτό τους και μεταξύ άλλων και ένας Γάλλος υπήκος. Είμαστε πολιτικοί εκλεγμένοι που οφείλουμε να καταδικάζουμε τη θανατική ποινή, όπως είπατε κι εσείς, γιατί την απαγορεύει η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε εκλεγμένοι πολιτικοί υπεύθυνοι και άνθρωποι που καταγγέλουμε αυτό το μακάβριο σκηνικό που συνοδεύει την καταδίκη σε θάνατο των υπόπτων στην Ινδονησία αλλά και αλλού όπως υπενθυμίσατε κύριε Επίτροπε. Πιέζει ο χρόνος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εταίρος της Ινδονησίας. Το Νοέμβριο που μας πέρασε στη Τζακάρτα είχαμε διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδονησία υπογράψαμε με την Ινδονησία Συμφωνία Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης. Είμαστε στη διάθεση της Ινδονησίας ε, στα πλαίσια των ε, περιφερειακών μας ε, συμφωνιών για να βοηθήσουμε στα περιφερειακά προγράμματα με κονδύλια. Ζητάω λοιπόν από τους Ευρωπαίους υπεύθυνου. Κάποιοι μάλιστα είναι στην ε, Τζακάρδα σήμερα για να υποστηρίξουν τους Ευρωπαίους υπηκόους, να πάνε πιο μακριά, να μην αρκεστούν σε διπλωματικά διαβήματα και ευγενικά λόγια, που μέχρι τώρα δεν είχαν αποτέλεσμα, γιατί το θέμα αυτό είναι ζωτική σημασία σήμερα για τους Ευρωπαίους πολίτες που περιμένουν τη βοήθειά μας. Βασίζομαι σε εσά για να μεταφέρετε στις αρχές της Ινδονησίας ένα μήνυμα ε, δυνατό, έντονο, που δεν παραβιάζει το δικαίωμά τους να καταπολεμήσουν τα ναρκωτικά, ούτε η ανάμειξη. Αλλά αυτό που κάνει σήμερα η Ινδονησιακή ε, δικαιοσύνη είναι κάτι σε βάρος ενός Γάλλου πολίτη που πρέπει να υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστούμε, συνάδελφε Νταζό. Ένα διαδικαστικό έχουμε τώρα στον τον Αλφάρνοτ. Yes, Mr. President. Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω από, από το άρθρο 162 υπό το σημείο 6 πώς ακυρώνεται το Catch the Eye γιατί αναφέρεται ότι θα δίδεται ο χρόνος αυτός. Θα ήθελα να μιλήσω για μια κυρία στην ε, περιφερειά μου που είναι προγραμματίζεται, έχει κάτι έχουν απαγγελθεί για ε, κατηγορίε κατηγορίες και μπορεί να καταδικαστεί σε θάνατο. Έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Θέλω να θέσω λοιπόν το θέμα αυτό. Συνάδελφε Άρνοντ, έχουμε κανόνε, λέει ο πρόεδρο. Οι κανόνε προβλέπουν ότι εδώ γίνεται μία συζήτηση Έκτακτη φύσεω και συμφωνήθηκε να μην υπάρξει διαδικασία ΚΑΣΤΙΑΙ και να μην υπάρξει και μπλε κάρτα. Και ε, επίση ο κανονισμό προβλέπει ότι το διαδικαστικό έχει να κάνει με το διαδικαστικό, όχι με θέματα περιεχομένου. Και σε κάθε περίπτωση στο μέλλον θα σα θερήσω το λόγο πολύ πιο γρήγορα. Όχι, λυπάμαι, δεν έχετε το λόγο. Το λόγο έχει ο συνάδελφο Μαρτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια μεγάλη χώρα μεγάλη δύναμη, αλλά πέρα από τη δύναμή της, λόγω των ιδεών της, της γενοδορίας που έχει αποδειχθεί επανειλημμένος κατά την ιστορία της. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, η δήλωση αυτή δεν είναι δικιά μου. Ο Ρομπέρ Βανταντέρ την έχει υπογράψει όταν ήταν υπουργό δικαιοσύνη στη Γαλλία το 1980. Αν λοιπόν αυτό το ίδιο μήνυμα που θέλω να στείλω εκ μέρους μας, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Ινδοσιακές Αρχές, ακουστεί, θα ήταν καλό. Ναι, Κύριε Πρόεδρε, το μπορείτε να είσαστε μεγάλος. Η γενοδορία σας πρέπει να φανεί στον κόσμο και η δύναμή σας να βοηθήσει τη ζωή. Πρέπει να στείλουμε και στους πολίτες της Ινδονησίας αλλά και του υπόλοιπου κόσμου ένα ισχυρό μήνυμα. Κανείς δεν αμφιβάλλει για την ε, επιθυμία σας να καταργήσετε τα ναρκωτικά, να τα παλύψετε. Είναι ένας βασιλιανό ε, Αυστραλιανή, Ινδονήσιος κλπ. Όλοι μαζί είμαστε κατά της ε, καταδίκης σε θάνατο. Όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν το θάνατο. Πρόκειται για βασανιστήρια ψυχολογικά που φύστανται οι καταδικασμένοι σε θάνατο και οι οικογένειές τους. Ξέρετε τι σημαίνει να περιμένει κανείς μια δίκη που δεν είναι στην πραγματικότητα δίκη. Χρειάζεται ανθρωπισμός. Όλα αυτά τα χρόνια περιμένουν οι άνθρωποι δικαιοσύνη, δίκαια και θέλουν την αλήθεια. Όλα αυτά είναι χρόνος αφόρητος για τους ανθρώπους αυτούς όταν κάθε προσφυγή απορρίπτεται από την Ινδονησιακή δικαιοσύνη και το μόνο που μένει είναι ο παγωμένος θάνατος. Στον ε, Σεζαταλή που είναι Γάλλος υπήκος από το δικό μου το διαμέρισμα θέλω να πω το εξής. Ο Σερ ζει 10 χρόνια τώρα αυτό το βασανιστήριο υποφέρει ψυχικά και νιώθει ένοχος που εξακολουθεί και βρίσκεται στη ζωή. Όχι σε. δεν είσαι ένοχος, δεν είσαι ένοχος που θέλεις να ζήσεις, δεν είσαι ένοχος που θέλεις δικαιοσύνη, δεν είσαι ένοχος που θέλεις να ξαναδείς τα τέσσερα παιδιά σου, δεν είσαι ένοχος που υποφέρεις εσύ και η δική του σε σκέφτομαι, Σέρ, τη σύζυγό σου, τα παιδιά σου και την οικογένειά σου που σε περιμένουν. Κράτα γερά, Σέρς. Η Γαλλία σε υποστηρίζει, η Ευρώπη πρέπει να σε υποστηρίζει και αυτό ακριβώ το μήνυμα είναι που θέλω να στείλω. Ζαν Ζωρέ έλεγε ότι η καταδίκη σε θάνατον είναι αντίθετη σε αυτά που και εδώ και 10.000 χρόνια σκέφτεται η ανθρωπότητα. Στην Ευρώπη λοιπόν, όπω και αλλού στον κόσμο ολόκληρο, κανένα άνθρωπο κόβεται το μικρόφωνο του ομιλητή σας ευχαριστώ και τώρα το λέγω έχει ο συνάδελφος Δεμές Μάκερ για 1,5 λεπτό. Η εκτέλεση των οκτώ καταδικασμένων στις αρχές της, ε, του μήνα προκάλεσε να σε όλο τον κόσμο. Και η ομάδα του ECR λοιπόν συμμερίζεται αυτή την αγανάκτηση. Α, για λόγους αρχής και βάσει του άρθρου 2 στο Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλους μας και κυρίως εμάς τους Ευρωπαίους ηγέτες που φαίνεται έχουν χάσει ε, την, ε, το τι σημαίνει, έχουν ξεχάσει τι σημαίνει το ότι δεν έχουμε δικαίωμα να καταδικάσουμε σε θάνατο, επαναλαμβάνω το εξή. Δικαίωμα στη ζωή. Ότι όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή και κανεί δεν μπορεί να καταδικαστεί σε θάνατο και να εκτελεστεί ε, σεβόμαστε την κυριαρχία της Ινδονησίας και την επικυριαρχία της. Είναι ένα σύγχρονο κράτος με εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη, αλλά η ηθική πτυχή δεν θα πρέπει να παραμεληθεί. Και αυτό ε, εκφράζεται σε πολλούς δομείς, στην ελευθερία του τύπου, ελευθερία εκφράσης, μέχρι το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η εκτέλεση της ανθικής ποινής παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, κατάλληλη ε, ανταπόκριση θα ήταν να μεταφραστεί σε ισόβια κάθριξη η καταδίκη αυτή. Τους αξίζει η φυλακή, αλλά όχι να δολοφονηθούν. Και εκ του ονόματος της ομάδας ECR, ε, οι συνάδελφοι Charles Stanox και εγώ ε, γράψαμε μια αποστολή προς τις αρχές της Ινδονησίας, αλλά δεν ωφέλησε σε τίποτε. Ελπίζω ότι, να ότι θα ακούσει σήμερα η Ινδονησία το μήνυμά μας. Σταματήστε σας παρακαλώ με τις εκτελέσεις σας ευχαριστούμε και τώρα για δύο λεπτά το λόγο έχει συνάδελφος Χάκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταδικάζουμε αυτές τις βίες εκτελέσεις με εκτελεστικό απόσπασμα 8 ανθρώπων στην Ινδονησία και 7 από αυτού δεν ήταν καν πολίτε τη Ινδονησία. Και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Αυστραλία απέθυναν σε εκκλήσει τι αρχέ να μην προχωρήσουν στην πραγματοποίηση των εκτελέσεων. Προσέφερε και βοήθεια όμω στι αρχέ, στι Ινδονησιακέ αρχέ, ε, για να αντιμετωπίσουν το αθρεμπόριο των ναρκωτικών. Η, τιμω, η τιμωρία επιβάλλεται στου καταδικασμένους μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινο τρόπο και μετά από δίκαιη ε, δίκαιη και θέλουμε να σταματήσουν όλες οι εκκρεμούσεις εκτελέσεις στην Ινδονησία. Αλλά είναι αρκετά ειρωνικό συνάδελφοι και ε, επέσχυντο όταν ακούσαμε τα φρικτά νέα για τις εκτελέσεις στην Ινδονησία ο Βίκτορ Ορμπάν το οποίο παραμένει το κόμμα μέλος του ΕΛΚ πρότεινε η θανατική ποινή να επανέλθει στην Ουγγαρία. Τέτοιε προτάσει είναι ε, εντελώ απαραδέξεις. Όπω γνωρίζει ο κ. Ορμπάν η θανατική ποινή απαγορεύεται στην Ευρώπη και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό καθώς και για τις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλουμε για τη λήξη της θανατικής ποινή, να περιοριστεί η εφαρμογή αυτής και να παγώσουν όλες οι χώρες σε αυτή την απάνθρωπη τιμωρία. Έχουμε βάλει τον πύχη ψηλά σαν Ευρώπη και θέλουμε να αυξάνεται το ύψος σαν φιλελεύθερες δημοκρατίες και θα ενισχυθεί η φωνή των δημοκρατιών απευθύνοντας εκκλήσεις όπως είναι η Ινδονησία σε χώρες αυτές αν είχαμε και τις ΕΠΑ στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν και η ε, έθεταν εκτός νόμου τη θανατική ποινή. Θα πρέπει να συνεχίσουμε παγκοσμίες προσπάθειες συνεργαζόμενοι με κυβερνήσεις, κοινωνίες των πολιτών, οργανώσεις αυτών να εξασφαλίσουμε ότι η θανατική ποινή σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν. Σα ευχαριστώ συνάδελφε Σάκη και τώρα για δύο λεπτά το λέγω έχει Άλφο Μπριζιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες που συμφώνησαν να συζητήσουμε στην ημερήσια διάταξη μετά από έτοιμα της ΓΚΟΕ το θέμα αυτό, για να καταπολεμήσουμε τη θανατική ποινή. Την Τρίτη το βράδυ, 8 άτομα εκτελέστηκαν ένα Ινδονήσιο και 7 ξένοι. 14 εκτελέσει από την αρχή τη χρονιά. Ενώ το 2014 δεν υπήρξε καμία, ενώ 5 μόνο το 2013 μετά από μια συμφωνία 5 ετών. Και στην Οδεονησή, όπω και αλλού, προσφεύγουμε κυρίω για τα ναρκωτικά στη θανατική ποινή. Για να αντιμετωπιστεί ένα έγκλημα, χρησιμοποιούμε ένα άλλο έγκλημα. Η προσφυγή σε αυτήν την ποινή, τη βάρβαρη, την επιβάλλουν πολλές φορές σε ξένους, σε μικρούς εγκληματίες που κάνουν τα βαποράκια. Λίγοι πραγματικοί βαρώνοι των ναρκωτικών περιμένουν τη θανατική ποινή στους διαδρόμους του θανάτου των Ινδονησιακών φυλακών. Στις 12 Μαΐου άλλοι δύο Αυστραλιανοί περιμένουν το απόσπασμα. Έχουμε 57 άλλους, από τους οποίους 27 είναι ξένοι, που έχουν καταδικαστεί σε... για ναρκωτικά. Τέσσερις Ευρωπαίοι. Ένας από αυτούς, 51 ετών, ο οποίος δούλευε σε ένα εργαστήριο της Ινδονησίας, υποστηρίζει ότι δεν ήξερε ότι το εργαστήριο στο οποίο δούλευε φτιαχνόταν η έκσταση. Ζήτησε να ξαναγίνει η δίκη του. Δεν απειλείται άμεσα η ζωή του. Το ίδιο και για έναν Κινέζο που έχει καταδικαστεί σε θάνατο για το ίδιο ακριβώς. Πολλές μαρτυρίες και αστυνομικών λένε ότι δεν φταίνε. Δεν έχουν ληφθεί όμως υπόψη. Ο πρόεδρος είναι ένας εθνικιστικής στην Ινδονησία που θέλει να δώσει την εικόνα κάποιου που δεν πιέζεται από το εξωτερικό με τίποτα. Το έχει κάνει όμως για μια γυναίκα από, την, από τις Φιλιππίνες. Η συζήτηση και στο Τζακάρτα Γκλόμπου, που είναι η κύρια Ινδονησιακή εφημερίδα συνεχίζεται και αναρωτιέται η εφημερίδα ποιο είναι το τίμημα για την Ινδονησία τελικά, τι εικόνα δίνει προς τα έξω η χώρα με τις θανατικές αυτές καταδίκες. Η Ινδονησία, Ηνωμένε Πολιτείε, Ευρώπη, ναι, ο Βίκτορ Ορμπάν πράγματι φαίνεται ότι είπε πως θέλει να ισχύσει και πάλι θανατική ποινή. Πρέπει να αντιδράσουμε όλοι μαζί και να συνεχίζουμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την αδελφέ Βερζιά και τώρα η συνάδελφος Λόχπιλερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν από δύο ημέρες στην Ινδονησία ε, εκτελέστηκαν οκτώ άνθρωποι. Η Ινδονησία το 2014 δεν έκανε καμία εκτέλεση, αλλά δυστυχώς φέτος έχουν γίνει ήδη 15 εκτελέσεις όλοι οι εκτελεστέντες ε, είχαν καταδικαστεί για λαθρεμπόριο ναρκωτικών παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διεθνές διατάξεις ε, όπου υπάρχει θεματική ποινή θα πρέπει να υπάρχει μόνο για τις πιο βαριές περιπτώσεις. Οι πρόσφατες λοιπόν εκτελέσεις στην Ινδονησία καταδεικνύουν ε, την έλλειψη σεβασμού των διεθνών προτύπων και διατάξεων για τη θεματική ποινή. Για παράδειγμα, ένας από τους κρατούμενους δεν είχε πρόσβαση σωστή σε διερμηνή, σε διερμηνία όταν κατούντων. Ένας ε, από τους κρατούμενους διαγνώστηκε με σχιζοφρέ... ως σχιζοφρονής παρά το γεγονός ότι απαγορεύεται σύμφωνα με διεθνή, διεθνή διατάξεις η εκτέλεση, η θανατική ποινή σε άτομα που έχουν πνευματικά προβλήματα δεν υπάρχει απόδειξη ότι η πίνη ποινή ε, αποτρέπει εγκλήματα. Και μία μελέτη του ΟΗΕ καταδεικνύει ότι δεν έχει, για παράδειγμα, η θανατική ποινή μεγαλύτερο αντίκτυπο αποτρεπτικό σε σχέση με την ισοβία κάθερξη. Ζητούμε λοιπόν από την ε, κυβέρνηση της Ινδονησίας να αναστείλει τις υπόλοιπες ε, προγραμματιζόμενες εκτελέσεις και να κάνει ένα μνημόνιο σε ό,τι αφορά να σταματήσει τις ε, εκτελέσεις. Και έτσι μπορεί η Ινδονησία να, θέσει ένα σημαντικό, να δώσει ένα σημαντικό μήνυμα και στις άλλες χώρες της περιοχής. Ευχαριστώ για δύο λεπτά τώρα. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Καστάλντο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, στο Σαμπαγκάν είναι ένα νησί και εκεί στην κοιλάδα του θανάτου συνονεύονται οι καταδικασμένοι με μεγάλη ασφάλεια φοράνε άσπρες φόρμες και είναι μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Μερούν να τους δέσουν τα μάτια, να καθίσουν, να γονατίσουν ή να είναι όρθιοι. Αυτή είναι, αυτός είναι ο ανθρωπισμός, η να ειναι ορθιοι αυτο ειναι αυτος ειναι ο ανθρωπισμος η ανθρωπια που τους δίνουν. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τις δίκες αλλά τη θανατική ποινή σαν κύρωση. Την καταδικάζω σαν Ιταλός, σαν Ευρωπαίος, αλλά πάνω απ' όλα σαν ανθρώπινο όν. Δεν υπάρχει εμπορικό συμφέρον που θα πρέπει να θυσιαστεί για μια συνεχή καταπολέμηση, για να καταπολεμηθεί θανατική ποινή και να τεθεί παρ... παρ ο κ. Κουρμάν έλεγε ότι είναι προφανές ότι εκείνοι που υποστηρίζουν τη θανατική ποινή σήμερα είναι πιο κοντά στους δολοφόνους από εκείνους που πολεμούν τη θανατική ποινή. Σας ευχαριστώ και στο τέλος ε, του γύρου αυτό το λόγο έχει πάλι ο Επιτρόπος Μίμητσα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Ήταν ε, πραγματικά ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων αυτών και σα ευχαριστώ για την σαφήνεια και την στοχοθέτηση των παρεμβάσεών σα. Θα ήθελα να σα βεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει απόλυτα δεσμευμένη στι επαφέ με την κυβέρνηση τη Ινδονησία, με του ακτιβιστέ και όλου του άλλου εμπλεκόμενου φορεί για να εργαστεί για την κατάργηση τη ε, θανατική ποινή στην Ινδονησία. Και θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα εργαλεία δηλώσεις, διαβήματα και διάλογο για να ακουστεί η φωνή μας, αλλά για να ακούσουμε και να κατανοήσουμε κάποια από τα εμπόδια στην αλλαγή, προκειμένου να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά. Καλούμε τις ε, αρχές και τον πρόεδρο της Αντωνησίας να αναστείλουν άμεσα την χρήση της αντικής ποινής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Και έτσι ολοκληρώθηκε η συζήτηση αυτή. Επόμενο